Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ένα διαδικαστικό υπό το άρθρο 11 τμήμα 3. Πέρυσι η διάσκεψη των Προέδρων διόρισε τον κύριο Γκίφερ Χόφστατ ως, Ευρωπαί... ως τον διαπραγματευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Brexit. Αλλά ο κύριος Φερχόφστατ επιπλέον έχει τέσσερις εξωτερικές θέσεις, κατέχει τέσσερις εξωτερικές θέσεις. Τρία εξ αυτές ε, αμείβονται με 5.000 ευρώ το μήνα και το κοινοβούλιο το πληρώνει πάνω από 10.000 ευρώ το μήνα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο κ. Φερχόφστατ είναι βεβαίως ένας άνθρωπος που διακρίνεται για την ακαιρεότητά του, την εντυμότητά του, αλλά πώς γίνεται ένας τέτοιος άνθρωπος ε, της ακυριότητας του κυρίου Φερχόφιστατ ε, με καθαρή συνείδηση να κληρώνει ε, όλες τις ευθύνες και τα καθήκοντα με όλες τις εξωτερικές του αυτές τις θέσεις ενώ παραμένει διαπραγματευτής του Κοινοβουλίου για το Brexit. Μήπως εγώ ζητώ λοιπόν να επανεξετάσουμε αυτόν τον διορισμό. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Πρόεδρε, αφού το Βρετανικό Κοινοβούλιο πέρασε το Brexit χτες το βράδυ και το άρθρο 50 θα τεθεί σε εφαρμογή πριν τα τέλη του μήνα, θα πρέπει να λάβουμε τις, τα μέτρα μας και εμείς. Αν ότι όποιο θέλει να καταστρέφει την Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει 260 επιδόματα χωρίς να δουλεύει καθόλου εδώ στο σώμα και στις επιτροπές. Εάν ε, ήταν σωστό, θα αρνούνταν τα προνόμια όσων θέλουν να παραμείνουν εντός της Ένωσης. Ευχαριστώ. Grazie, grazie Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την πρότασή σας, αλλά εδώ δεν θα συζητήσουμε το Brexit σε αυτή εδώ τη σύνοδο. Θα έχουμε μακρές και σημαντικές συζητήσεις για αυτό το θέμα και θα έλεγα να περάσουμε στις σημερινές μας εργασίες. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαν, να ρωτήσω μάλλον τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαν, αν η απουσία του αρμόδι, της αρμόδιας Επιτρόπου Πιανκόσκα για την εσωτερική ε, αγορά και του κ. Κατάινεν ε, για να στην διάρκεια της συζήτησης της οδηγίας περί ε, πυροβόλων όπλων ήταν η θελημένη. Εδώ το Κοινοβούλιο έχει περάσει ένα χρόνο λέγοντας στην Κομισιόν ότι δεν πρόκειται για την τρομοκρατική νομοθεσία. Ακριβώς λόγω της ελεύθερης κυκλοφορίας των, ε, προσώπων χρειάζεται ένα ελάχιστο κοινών κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν μας ακούτε και κάνετε, ε, ε, τόσο δυσχεραίνετε το έργο μας και δεν καταφέρνετε να μιλήσετε για αυτό το θέμα που μας απασχολεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος, η Άννα Γκόμες. Κύριε Πρόεδρε, Μια τραγωδία συνέβη πριν από δύο μέρες στην Αιθιοπία με, πάνω, με το θάνατο πάνω από 60 ανθρώπων, παιδιών και γυναικών κυρίως σε μια ε, σε κάποια χωματερή Και μάλιστα αυτό συνέβη σε μια χώρα που είναι μέγας δικαιούχος ε, κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από την ε, έκφραση της αλληλεγγύης μας με το, προς το λαό της Αιθιοπίας, θα έπρεπε να απαιτήσουμε η Κομισιόν να διερευνήσει ποιο είναι το επίπεδο κακής διαχείρισης, κακοδιαχείρισης και ε, στη χώρα αυτή, στην Αιθιοπία, όταν ο κόσμος χάνει τη ζωή του και βρίσκεται στο έλεος μιας απόλυτα αντιδημοκρατικής δικτατορίας. Σας ευχαριστώ. Έχω αποφασίσει να επιβάλλω κύρωση κατά του κυρίου Κόρβιν Μίκε. για τις παρατηρήσεις και δηλώσεις που έκανε σχετικά με τις γυναίκες κατά την Σύνοδο Ολομελίας της 1ης Μαρτίου του 2017 κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις αποκλήσεις αμοιβών μεταξύ των φίλων και με προεδρία γυναίκας αντιπροέδρου της κυρίας Γκέπχαρτ. Θεωρώ ότι οι δηλώσεις αυτές και παρατηρήσεις συνιστούν παραβίαση των αρχών που ορίζει το άρθρο 11 του εσωτερικού κανονισμού. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 166 του εσωτερικού κανονισμού και ε, λαμβανομένων υπόψη των γραπτών παρατηρήσεων που υπέβαλε ο κύριος Κορβιμίτ και αποφάσισα να επιβάλλω τις εξής κυρώσεις. Πρώτον, παρακράτηση των βουλευτικών αποζημιώσεων για περίοδο 30 ημερών. Δεύτερον, και με κάθε επιφύλαξη του δικαιώματο για συμμετοχή στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια, προσωρινή αναστολή από τη συμμετοχή όλων των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου για περίοδο 10 ημερών, αρχής γενομένης από σήμερα. Επιπλέον, ο κύριος Κόρβιν Μίκε δεν επιτρέπεται να εκπροσωπεί το κοινοβούλιο σε, το κοινοβούλιο σε ιαδήποτε διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, διακοινοβουλευτική διάσκεψη ή διοργανικό φόρουμ για περίοδο ενός έτους αρχής γενομένης από τη σήμερον. Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο βουλευτή. Και τώρα περνούμε στις ψηφοφορίες. Περνούμε τώρα στις ψηφοφορίες. Έκθεση Γκέρλινγκ.